Έχουμε πρώτη την ελευθερία τη έκφραση του Καζακστάν. Με συντάκτε γνωμοδοτήσεων που θα λάβουν πρώτο το λόγο και τους καλώ. Συγγνώμη, ε, δεν ομιλώ εκ μέρου τη ομάδα μου, ούτε και με και συντάκτη, λέει κυρία Ζητάνοκα. Επομένω, Μάλλον θα λάβω το λόγο αργότερα. Η πρόεδρος πολύ καλά. Για να δω τον κατάλογο. Εγώ σας βλέπω ως συντάκτη. Και για μετά δεν θα μπορώ να σας δώσω το λόγο. Λοιπόν, ή τώρα ή ποτέ. Καλώς, κοιτάξτε. Να μιλήσω λοιπόν ε, ως μέλος της αντιπροσωπείας για τη σχέση με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Εγώ θέλω έναν ισότιμο διάλογο σε συνθήκες αμοιβαίου σεβασμού με το Καζακστάν. που έχει πολύ μεγάλη σημασία στην περιοχή του και θέλω να διατυπώσω τα εξής ερωτήματα προς τους συναδέλφους εάν δεν εξετάζουν με σοβαρότητα την ε, αίτηση του Καζακστάν να καταστεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 17-18 και να του επιτρέψει αυτή τη συμμετοχή πώς μπορούμε εμείς να ε, κάνουμε μαθήματα στο Καζακστάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όταν εμείς κάνουμε τα ίδια και χειρότερα στην ίδια περιοχή μέτρα τα οποία λήφθησαν τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία, επί παραδείγματι, από ό,τι μα λέει και το Συμβούλιο τη Ευρώπη, έχουν οδηγήσει σε συστηματική υποβάθμιση των δικαιωμάτων του κράτου δικαίου, το, της ελευθερίας της έκφρασης των θεμελιωδών ελευθεριών. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε εξίσου να συζητήσουμε το κράτο δικαίου για, και την ανεξαρτησία των μέσων μαζική ενημέρωση στην Πολωνία. Στην Λετωνία, την πατρίδα μου, υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση μια σειρά νέων διατάξεων στο ποιδικό κώδικα, που προβλέπουν ποινές φυλάκισης ακόμη και για μη βίαιη δράση κατά της κυβέρνησης και συνεργασία με ξένες οργανώσεις εις βάρος των συμφερόντων ασφαλείας της χώρας. Εγώ προσωπικώς καταδικάζω απερίφραστα κάθε παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης ανά τον κόσμο. Πρέπει να αγωνιστούμε για αυτές τις ελευθερίες όλοι μαζί και όχι ο ένας απέναντι στον άλλον. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Εγώ καταλαβαίνω το πρόβλημα γιατί σας είχαμε προβλέψει για τη συζήτηση τώρα. Ο κύριος Κορράου. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στο Καζακστάν επηρεάζει τις εμπορικές μας σχέσεις. Οι μειονότητες υφίστανται ε, πολλές ενέργειες καταστολής από πλευράς των αστυνομικών αρχών, γίνονται αυθαίρετα παράνομες κρατήσεις, χρησιμοποιείται συστηματικά, ε, χρησιμοποιούνται τα βασανιστήρια, περιορίζεται η ελευθερία συγκέντρωσης, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία τύπου. Υπάρχει μια μάλιστα πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που περιορίζει ακόμα περισσότερο την ελευθερία έκφρασης και φύγει φυσικά αυτούς που είναι στην αντιπολίτευση και τους δημοσιογράφους. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι κυρώσει, θα πρέπει να ληφθούν εις βάρος αυτών των ενεργειών. Ίσως εδώ θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν συμφέροντα που εμποδίζουν την λήψη μέτρων. Ο κύριος Τσαρνέσκι είναι ο επόμενος. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ξέρετε συνάδελφοι. Δεν θα μιλήσω όπω κυρία Τσαρόσκα για την κατάσταση στη Λετωνία. Εγώ θα μιλήσω για την κατάσταση στο Καζακστάν. Έχω επισκεφθεί τη χώρα αυτή 7 φορές στην, Αρμα, στην Αλμάτα πρώτα και μετά στην Αστάνα, δύο διαφορετικές πρωτεύουσες. 2.000 χιλιόμετρα διένυσα με τα αυτοκίνητα διέστησε ολόκληρο το Καζακστάν και θεωρώ ότι γνωρίζω αρκετά καλά τη χώρα. Και πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο όταν ε, λαμβάνουμε το λόγο να μιλούμε για πράγματα που γνωρίζουμε. Γνωρίζω λοιπόν αρκετά καλά το Καζακστάν. Η κατάσταση στην περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερη. Ολόκληρο το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπινών δικαιωμάτων είναι αντιληπτό σε όρους διαφορετικούς από ό,τι το εννοούμε εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό και υποστηρίζω το ψήφισμα. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι σημαντικά τα θέματα. Ο κύριος Κέλαμα έχει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Χάν, ανησυχούμε βαθύτατα για την ελευθερία της έκφρασης στο Καζαχστάν η πρόσφατη υπογραφή της ενισχυμένης Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας βεβαίως είναι ένα θετικό βήμα για την ενίσχυση των σχέσεων, αλλά οι σχέσεις πρέπει να στηρίζονται σε κοινέ αξίες και δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Και δεν, σας κάνουμε, και δεν κάνουμε διδάγματα σε, σε, σε έναν εταίρο, απλώς μοιραζόμαστε με τον τρόπο αυτό τις ίδιες αξίες. Υπάρχουν ανησυχίες λοιπόν και φωνές επίκρισης που φημώνονται με την υπογραφή τον προηγούμενο Δεκέμβριο αυτή τη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία, βλέπουμε να οξύνονται οι επιθέσει βάρο των δημοσιογράφων. Η Τελιένοβα και η Κασλόβα με την ιστοσελίδα του ε, που έκλεισε κατηγορήθηκαν για την, ε, και συνελήφθησαν για διάδοση ψευδών ειδήσεων. Ο Κασλόφ, άλλοι δημοσιογράφοι όπως Λούκες, Μάτοι, Μαμπετάλιν, Πιέλοκ έχουν μπει στο στόχαστρο. Μπορεί να σας φαίνονται μακρινά, μακρινός ο ήχος των ονομάτων τους και όχι πολύ εγγύης, αλλά πρέπει να τους δείξουμε αλληλεγγύη, μια πραγματική αλληλεγγύη προς τους δημοκρατικούς πολίτες. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. ΠΑΕΤ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα δημοσιογράφοι και μπλόγγερ να έχουν επανειλημμένα συλληφθεί, να έχουν υποστεί πιέσει και απειλέ από τι αρχέ μόνο και μόνο για την εκδήλωση των απόψεών του. Ε, υπάρχουν πολλέ πιέσει και σε σχέση με τι ε, δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Πρέπει λοιπόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών να είναι σε θέση να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους χωρίς φόβο παρενοχλήσεων και πιέσεων. Πρέπει να βελτιωθούν οι σχέσεις ε, των ανθρωπινών δικαιωμάτων, πρέπει η συμβατική και εταιρική σχέση με το Καζακστάν να οδηγεί σε βελτίωση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και του σεβασμού του κράτους δικαίου. Χαίρομαι βεβαίως γιατί το Καζακστάν έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Είναι σημαντικό εξίσου όμως το Καζακστάν να υλοποιήσει τις διεθνείς του υποχρεώσεις σε άλλες σφαίρες για το κράτος δικαίου, για την εξασφάλιση δικονομικών εγγυήσεων για την προστασία των επενδύσεων των επενδυτών από το εξωτερικό. Και σας ευχαριστώ πολύ. Σάντσες Κάλντεντε, παρακαλώ, αυτό το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Καζακστάν μετά από ε, την Σοβιετική εποχή είναι πλέον χάρη στις, ε, στα πετρελαία πετρελαϊκά το κοιτάζουμε τα πιο πλούσια από τις ε, χώρες αυτού του μπλοκ. Δυστυχώς όμως υπάρχει επιδείνωση των συνθήκων, διαφθορά, τα επιχειρηματικά και τα πολιτικά συμφέροντα είναι συγκεχημένα, υπάρχει απολυταρχικό καθεστώς, ε, υπάρχει ε, καταδίκη και καταδίωξη όλων όσων ασκούν κριτική, bloggers, δημοσιογράφοι κτλ. Επίσης παραβιάζονται συστηματικά οι συνθήκες ε, εργασίας, τέλονται συνδικαλιστικές ελευθερίες ελευθερίες. Είναι πολύ άσχημο αυτό το πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα αναθεωρεί τη στρατηγική τη ε, για την κεντρική Ασική, ε, Ασία με βάση μόνο πολιτικού και οικονομικού στόχου, χωρί να λαμβάνει υπόψη για μια ακόμη φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι κατεπίγον αρχή να μα απασχολεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη εκείνα που θεωρούμε εταίρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να έχει σχέσεις με ανθρώπους που παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο έχει το λόγο. E Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συλλήψεις δημοσιογράφων και μπλόγκερ τον προηγούμενο Δεκέμβριο, λίγες μέρες πριν από την υπογραφή της ενισχυμένης εταιρικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ένωση και το Καζακστάν, Θυμίζω ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει ξεκάθαρες ρήτρε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι ανησυχητικό μήνυμα. Πέρα από τις πρόσφατες περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνονται ε, στο ψήφισμα φαίνεται ότι και οι αρχές του Καζακστάν προσπαθούν να φημώσουν ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης ε, τα οποία έφυγαν από τη χώρα και εκπέμπουν από το εξωτερικό όπως το Ρεσπούμπλικα. Είναι πολύ ανησυχητική η χρήση του άρθρου του κώδικα του ποινικού που χρησιμοποιείται εις βάρος των συγκεκριμένων ανθρώπων που ασκούν κριτική στις αρχές ε, χωρίς κανένα άλλο επιχείρημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τους συντάκτες. Περνάμε τώρα στους ε, εκπροσώπους ε, ε, των ομάδων από το ΕΛΚΟ, κύριος ε, Πρόσπισιλ, κατάρχας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, τους συντάκτες δηλαδή, που είπαν πολύ σωστά ότι εδώ συζητούμε την ελευθερία λόγου, τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν, που έχει υπογράψει στρατηγική συμφωνία. επομένως πρέπει να μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τις βασικές ελευθερίες και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα αυτή η χώρα. Ελευθερία του συνέρχεστε, συνεταιρίζεστε, δημόσια έκφραση κτλ. Όλα αυτά είναι ακόμα πιο σημαντικά αν ληφθούν υπόψη οι επικείμενε εκλογές στο Καζακστάν σε λίγε ημέρε έχουμε πάρα πολύ γρήγορες ε, κοινοβουλευτικές εκλογές. Πρέπει να τις παρακολουθήσουμε. Πρέπει να δούμε γίνονται σεβαστή η ε, αρχή της καθολικής μυστικής ψηφοφορίας. Έχει περιγραφεί επίσης διεξοδικά η καταπίεση απέναντι σε ε, αντιπολιτευόμενους, σε δημοσιογράφους, σε bloggers. Θέλουμε να έχουμε αυτό το στρατηγικό εταίρο το Καζακστάν, αλλά για να έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση θα πρέπει να απελευθερωθούν ε, στη χώρα αυτή όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι οι bloggers που κρατούνται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Λεπρόεδρε. Λαουρίστε την επόμενη ομιλήτρια, παρακαλώ μισή λεπτό έχετε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη. Οι Σοσιαλδημοκράτε, ε, μπορεί να λένε εκ μέρου μα ή όχι ότι ναι μεν γίνονται ε, κάποιες προσπάθειες που είναι σημαντικές και τις ε, υποστηρίζουμε, αλλά από την άλλη πλευρά το Καζακστάν θα πρέπει να τηρήσει αυστηρά όλες τις δεσμεύσεις του. Υπάρχουν όμως, ε, βλέπουμε αντιφάσεις εδώ. Το Καζακστάν στρέφεται ε, με σφοδρότητα κατά οποιονδήποτε αντιφρονούντων. Και μάλιστα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ με καθεστώς ε, πρόσφυγα. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν φύγει από τη χώρα. Ελπίζουμε ότι σε αυτή τη φάση που σίγουρα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε για αυτή τη συμφωνία των συναλλαγών, αλλά να κοιτάξουμε και το κατά πόσον το Καζακστάν φέρει σε πέρας και τις δικές του υποχρεώσεις, ε, εξασφαλίζει τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται όχι μόνο από τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών, αλλά και από το ίδιο το Σύνταγμα του Καζακστάν. Στηρίζω λοιπόν θερμά αυτό το ψήφισμα και καλό όλα τα κράτη-μέλη να εξετάσουν ε, το τι συμβαίνει στο Καζακστάν για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με άσκηση πιέσεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Κούσουκ, επόμενος ομιλητής, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε πίτρο Χάν, αγαπητοί συνάδελφοι όπως και οι υπόλοιπες ε, χώρες περιοχής ε, έτσι και εγώ πιστεύω ότι είναι προ... πλούσια η ιστορία αυτής της πρώην Σοβιετικής χώρας που ήταν η πρώτη χώρα ε, από την Κεντρική Ασία η οποία ε, συνήψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε κοινά project, κοινά σχέδια. Εδώ και 25 χρόνια αναζητά τη δημοκρατική της ταυτότητα η χώρα αυτή. Παρά το αυτό το πολιτικό σύστημα μοιάζει περισσότερο με ολιγαρχία τα τελευταία χρόνια. Οι δημοκρατικές αρχές καταπατώνται. Οι bloggers, οι δημοσιογράφοι στερούνται ε, της ελευθερίας τους. Για ποιο λόγο, γιατί πολύ απλά προβαίνουν σε ενέργειες για την άσκηση της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας λόγου. Καλό τις αρχές του Καζακστάν να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στη διεθνή κοινότητα και στο πλαίσιο της ΟΑΣΕ. Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, αλλά και πολίτες ε, που κρατούν φλεξ πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Φουντζούλησα. Τη δέχεστε? Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, όπω ξέρετε τώρα η Συμφωνία Εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Καζακστάν δεν έχει ακόμα ε, κυρωθεί από όλα τα κοινοβούλια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένη κατάσταση λοιπόν δεν νομίζετε ότι θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προ ορισμένα κοινοβούλια ε, κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβραδύνουν τη δικασία κυρώσου, έτσι ώστε να περιμένουμε να τηρηθούν από το Καζακστάν και οι ε, εκκλήσει που έχουμε διατυπώσει τι συστάσει για την ελευθερία τη έκφραση και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φουτζούλητσα για την ερώτησή σα, βεβαίω και συμφωνώ απολύτω μαζί σα Απολύτω. το Καζακστάν οφείλει να κάνει σεβαστέ όλε τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Κάθε δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης. Μόνο μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε το διάλογο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ο κύριος Ζαριανόπουλος έχει το λόγο, μία εγγεγραμμένος βουλευτής. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποκαλύπτεται ποια είναι η δίθεν δημοκρατία και ελευθερία που επιβλήθηκε στους λαούς της. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την κρατική βία της κυβέρνησης του Καζαχστάν, την καταστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και λαϊκών ελευθεριών, του ταξικού εργατικού κινήματος και των κομμουνιστών με την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Καζαχστάν η έκθεση αποσιωπά αυτά τα γεγονότα η κοινή έκθεση όλων των πολιτικών ομάδων. δεν αναφέρει κουβέντα για τη δολοφονική επίθεση της αστυνομίας στους απεργούς διαδηλωτές της πόλης ζαναοζέν το θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων από αυτούς το πογκρόμ διώξεων κατά δεκάδων άλλων αγωνιστών. ούτε αναφέρει τίποτα για τον νόμο για ασφυκτικό έλεγχο των εργατικών σωματείων. είναι υποκριτική και επιλεκτική η δίθεν ανησυχία τη ευρωπαϊκής ένωσης και του κοινοβουλίου καθώ ανάλογα μέτρα εφαρμόζονται και σε κράτη μέλη τη με την βούλα αυτών των οργανισμών. εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στους κομμουνιστές και το ταξικό κίνημα του καζαχστάν κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές του καζαχστάν. Σας ευχαριστώ. Κύριε ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Όλοι μας εδώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι όρος εκτελώνου άνευ ε, για να κάνει καλά τη δουλειά του οποιοδήποτε και πάνω απ' όλα ο δημοσιογράφος. Η ελευθερία στην ανταλλαγή απόψεων ε, είναι δικαίωμα δημοκρατικό. Δεν μπορεί κανείς να το περιορίσει, μπορεί κανείς να εμποδίσει την κυκλοφορία πληροφοριών, αλλά δεν μπορεί να την αποτρέψει. Και δεν είναι δυνατόν να διαδίδονται άλλου τύπου ισχυρισμοί και κατηγορίες προκειμένου να φημωθεί η ελευθερία του τύπου Φερρυπίν, κατηγορίες για άλλα θρεμπόριο ε, ναρκωτικών και διακίνηση παρανομών προϊόντων. Εγώ επιμένω για το 10D του προημίου μας. Η κυρία Κόσλουβα ε, κατηγορείται για εγκλήματα που ε, επισύρουν ποινίως και 7 ετών και δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε σε αυτό. Πρέπει να υπερασπιστούμε όλους αυτούς ε, που αγωνίζονται για την ελευθερία του στο Καζακστάν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά η κατάσταση με την ελευθερία έκφραση στο Καζακστάν ε, πόρο απέχει του να είναι ιδανική. Πολλά πρέπει να γίνουν και από την κυβέρνηση της χώρας αλλά και από την ε, κοινωνία εν γέννη. Πριν γίνω βουλευτής, ήμουν δημοσιογράφος, γνωρίζω πολλούς bloggers από το Καζακστάν, έχω συνεργαστεί μαζί τους, ε, τους είχα δώσει φωνή, τους είχα δώσει βήμα στη χώρα μου που δεν είχαν ε, την ευκαιρία να μιλήσουν στη δική, στη δική τους χώρα. Όμως, να πω και κάτι ακόμη. Μπορούμε να κάνουμε μαθήματα στο Καζακστάν όταν βλέπουμε τι γίνεται εδώ, στη χώρα μου, τη Λετωνία. Ο Μαξίμ Κοτέλοφ επειδή έγραψε στο διαδίκτυο ένα ε, αστείο για τη Λετωνία ότι τα έχει κάνει πλακάκια με τη Ρωσία ε, μπήκε 6 μήνες φυλακή ότι παραβίασε την ελευθερία έκφραση τελικά. Κύριε Μάνκη, ήσασταν ο τελευταίο ομιλητή και περνάμε τώρα στη διαδικασία προσέλκυση προσοχή ε, του Πρόεδρου με πρώτο τον κύριο Ταγιάννη. Αντώνιο, you have the floor. for the Ναι, ναι, έχουμε περάσει την επόμενη συζήτηση. Ή μάλλον ο κύριος Κούκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Καζακστάν είναι η πρώτη χώρα στην Κεντρική Ασία που υπέγραψε μια συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμπληρώνει τις προσπάθειες που έκανε η χώρα αυτή στον τομέα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Παρά τη στενή σχέση που έχουμε με το Καζακστάν, πρέπει εμείς να τονίσουμε την αυξανόμενη πίεση εις βάρος των ανεξάρτητων ΜΜΕ και επίσης και εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα καταστολής από πλευράς των αρχών. Ακόμα και η μάχη κατά της τρομοκρατίας δεν πρέπει να επιτρέπει τέτοια μέτρα ιδιαίτερα ε, στα πλαίσια μιας προεκλογικής περίοδου που πρέπει να αφήσει τους πολίτες να πάρουν μόνοι τις ελεύθερες αποφάσεις τους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω λοιπόν επίσης και τη μεγάλη σημασία που έχουν εδώ οι συστάσεις του ΟΑΣΕ. Ο κύριος Καπούτο. Eh, Κοιτάξτε, οι κάρτες αυτές τις σηκώνετε τόσο γρήγορα που δεν ξέρω για ποια συζήτηση σηκώνετε τις κάρτες. Περιμένετε λοιπόν σας παρακαλώ να κλείσει η συζήτηση. Ο κύριος Μαριάς, για ποιο θέμα έχετε το λόγο. Η οικονομία στο Καζακστάν έχει πληγεί σοβαρά από την πτώση της τιμής του πετρελαίου το εθνικό νόμισμα έχει χάσει τη μισή του αξία από το περασμένο καλοκαίρι και όλα δείχνουν ότι η κρίση θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του. 2016. χιλιάδες σε αυτές τις συνθήκες σκληρής πλέον οικονομικής κρίσης εκφράζεται η δυσαρέσκεια του λαού. πρέπει λοιπόν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων ιδίως του ρωσικού στοιχείου όπως επίσης και η βούληση του λαού του Καζακστάν. όμως το καθεστώς φημώνει την ελευθερία τύπου τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών παραβιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συλλογικές ελευθερίες. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να στείλει ένα αποφασιστικό μήνυμα στο καζακστάν το οποίο αποτελεί σημαντικό εμπορικό εταίρο της ένωσης. στην κεντρική ασία θα πρέπει να υπάρξει σταθερότητα και ανάπτυξη. αυτό όμως περνάει από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ειρηνική συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων. ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε αγαπητέ συνάδελφοι. Καστέλη, εσείς για αυτή τη συζήτηση θέλετε το λόγο ή όχι. Ο συνήθως, ε, καλούμεθα να σχολιάσουμε μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανιστήριων, άρνησης ε, της ελευθερίας έκφρασης ε, και μέσων ενημέρωσης ε, τα οποία ελέγχονται για λόγους εθνικής ασφαλείας από τις κρατικές υπηρεσίες. Οι δημοσιογράφοι υφίστανται διώξεις όταν προσπαθούν να κάνουν την δουλειά τους. Το ίδιο έπαθε και η εφημερίδα Ντάμπολ τον προηγούμενο Ιούνιο Επίσης ε, μπλοκάρεται η πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που θεωρούνται απειλητικές για την κυβέρνηση χωρίς καμία δικαστική απόφαση. Επίσης ε, το νέο άρθρο στον ποινικό κώδικα του 2015 για την προτροπή στην διχόνοια είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή είναι η κατάσταση στο Καζακστάν. Μην χρησιμοποιείτε παρακαλώ δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μην εγκαταλείπετε τα ανθρώπινα δικαιώματα μόνο και μόνο για λίγα βαρέλια πετρελαίου. κύριος Πότσακ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα συνεχίσω μετά από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Καστάλντο. Ο νέος ποινικό κώδικας μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ο συνάδελφος ε, ε, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Ο περιορισμός ε, της ελευθερίας συγκέντρωσης, δημιουργούνται προβλήματα στους κατοίκους του Καζακστάν, δεν μπορούν να διαδηλώνουν, δεν μπορούν να συνέρχονται. Νομίζω λοιπόν ότι η ελευθερία επίσης του τύπου είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Οι προεδρικές εκλογές δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν ακόμα και οι εκπρόσωποι, οι υποψήφοι μάλλον για πρόεδροι της αντιπολίτευσης λέγουν ότι καλύτερος από όλους είναι ο Ναζαρμπάγεφ. Ε, αυτό τώρα δεν ανταποκρίνεται ε, στους κανόνες της δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνει η συζήτηση ε, και θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χάν εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Η ελευθερία της έκφραση θα πρέπει να ε, εξασφαλίζεται από το Σύνταγμα του Καζακστάν και η διεθνή διάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και τι διεθνεί βεβαίω δεσμεύσει που έχει αναλάβει το Καζακστάν. Αυτά είναι προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ήταν στην πρώτη γραμμή των εκκλήσεων για τη βελτίωση τη κατάσταση και συνεχίζει να εγείρει ζητήματα σχετικά με την ελευθερία τη έκφραση τη διμερή σχέση με το Καζακστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ανησυχία για τις εντυνόμενες πιέσεις έναντι του ανεξάρτητου τύπου. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει αρκετά ε, έντυπα ή έχουν ε, επιβληθεί δυσανάλογα βαριά πρόστιμα εις τους. Αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με τις δημοσιεύσεις και τις συγκεκριμένες πιέσεις προς τα έντυπα αυτά, αλλά και προς ε, μία τάση να επιβληθεί στους λοιπούς ένα είδος αυτολογοκρισίας. διώξει έχουν ασκηθεί και κατά bloggers και για δηλώσεις που έχουν διατυπωθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων. Είδαμε με λύπη μας ότι ακόμα και εκείνοι που αποφυλακίστηκαν, αποφυλακίστηκαν με τον όρο, με περιοριστικούς όρους ε, ως προς την ελευθερία κινήσεών τους. Επίσης, ε, ε ποινικέ κυρώσεις για δυσφήμιση, για προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας είναι υπερβολικές. Καλούμε το Καζακστάν ιδιαίτερα να αναθεωρήσει το άρθρο 174 του ποινικού του κώδικα, το οποίο προβλέπει βαρύτατες κυρώσεις για μια σειρά από αδικήματα και το οποίο έχει αξιοποιηθεί επανελειμμένως εις βάρος ε, αγωνιστών ανθρωπινών δικαιωμάτων και μπλόγκερ. Η Ευρώπη διαρκώς διατυπώνει τις ανησυχίες της για την ελευθερία της έκφρασης ε, και, και τις εξελίξεις της κοινωνίας του Καζακστάν μέσα από τις συμφωνίες για εταιρική σχέση και συνεργασία. Κατά την επίσκεψη στην Αστάνα 21 Δεκεμβρίου πέρυσι για την υπογραφή της εν λόγω συνθήκης, η ύπατη εκπρόσωπος για τις, ε, για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα υπογράμμισε τη διάσταση των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παγίως επιδιώκει να στηρίξει την κοινωνία του Καζακστάν υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης και των δημοκρατικών ελευθεριών και των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο εταίρο ως προς την ε, αντιμετώπιση προς τα βελτίω αυτού του συγκεκριμένου ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε. Ανακοινώνω ότι έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος που θα ολοκληρώσουν την ε, συζήτηση και θα ψηφίσουμε στις 12 επ' αυτών. Το επόμενο θέμα στην μέση διάταξη, η Αίγυπτος και κυρίως η υπόθεση του Τζούλιου Ρετζένη. Θα δώσω το λόγο στους συντάκτες καταρχάς. Η κυρία Λόχπιλερ πρώτη. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση των δικαιωμάτων στην Αίγυπτο είναι δραματική και επιδεινώνεται διαρκώς. Οι Αιγυπτιακές αρχές καταστέλουν θεμελιώδεις ελευθερίες, ε, στην πραγματικότητα απαγορεύεται η αδίποτε δημόσια διαδήλωση, ασκούνται πιέσεις και απειλές ε, κατά ιδιωτών ή μέσω μαζικής ενημέρωσης. Οποιοςδήποτε διαφωνεί στην Αίγυπτο κινδυνεύει σοβαρά. Υπάρχουν αυθαίρετες κρατήσεις και προφυλακίσεις χωρίς καμία επαφή με τον ε, έξω κόσμο για εβδομάδες. Το Human Rights Watch έχει καταγράψει πάρα πολλές περιπτώσεις αγνοουμένων κρατουμένων που έχουν, και πολλών που έχουν βρεθεί νεκρύστερα από κράτηση από τις αρχές κράτησης δεν είναι φρικτές. Ε, πολλές είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων των κρατουμένων που δεν φτάνουν ποτέ ε, μέχρι τα δικαστήρια. Επισκέφθην την ε, Αίγυπτο πριν από μερικές εβδομάδες. Ήταν οι όπου είχε μόλις ανακαλυφθεί το νεκρό σώμα του ερευνητή Τζούλιο Ρετζένη και ήταν πολλοί μαζί με μένα οι οποίοι καταδίκασαν αυτές, ε, αυτήν και πολλές άλλες ε, παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να φταίνε μέλη του <clears throat> των ε, αρχών ασφαλείας και επιβολής της τάξης για την δολοφονία αυτή. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ε, λειτουργήσουν ικανοποιητικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο για να λειτουργήσει σωστά και το κράτος. δεν υπάρχει αυτό, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να ε, μείνουν συνένοχα και να επιτρέψουν αυτή την κατάσταση στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ, Μπέλτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πετρόπη, το δολοφονία του κυρίου Ρετζένη θα μπορούσε να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να δούμε τι προέκυψε από την κοινή έρευνα Αιγύπτου και Ιταλίας. Θα πρέπει να σταθμίσουμε και να μελετήσουμε καλά τα πορίσματα. Έχουν καταστραφεί επίσης πάρα πολλές εκκλησίες και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και την νομοθεσία περί Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί πιέσεις για κατάργηση του νόμου περί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει Τι πολιτική ασκεί τελικά απέναντι στην Αίγυπτο. Κοράου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Τζούλο Ρετζένι ήταν ένας Ευρωπαίος νέος ο οποίος ήθελε να βοηθήσει στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας, μιας ελεύθερης κοινωνίας. Η ερευνητική του δουλειά τον οδήγησε σε θέματα που δημιουργούσαν προβλήματα στις Αιγυπτιακές αρχές που ήθελαν να τα αποκρύψουν από την ε, δημόσια σκηνή. Αυτό οδήγησε λοιπόν τον Ρετζένι να βασανιστεί με βάρβαρο τρόπο και να δολοφονηθεί τελικά κάτω από συνθήκες άγνωστες ακόμα. Θα μπορούσε να είναι ο αδελφός μας, θα μπορούσε να είναι ο ανιψιός μας, θα μπορούσε να είναι ο φίλος μας. Παρά τους στενούς δεσμούς που έχουμε με την Αίγυπτο πρέπει να πάρουμε μια αποφασιστική θέση που ε, να ζητά να έχει φως στην ε, δολοφονία του Ρετζένη δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με τον ρόλο τον οποίο έπαιξαν οι δημόσιες αρχές. Βλέπουμε τη φωτογραφία του εδώ, την αφιερώνουμε στην οικογένειά του και στους φίλους του. Ζητάμε την αλήθεια για το Ρετζένι. Ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι θέλουμε την αλήθεια, θέλουμε τη δικαιοσύνη. Έθεσα το θέμα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την παρουσία της κυρίας Μογκερίνη η οποία αγνόησε την υπόθεση Ρετζένη. Δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτή. Ε, υπάρχουν ε, όλα σχεδόν οι πολιτικές ομάδες οι οποίες υπογράφουν ε, την συγκεκριμένη πρόταση. Εμείς έχουμε, θεωρούμε ότι είναι πολύ χαλαρή και θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να αυτολογοκρινόμεθα. Όταν η Αίγυπτος ήταν υπό την εξουσία του Μόρση και όταν ήταν στην εξουσία οι αδελφοί μουσουλμάνοι ε, τους έβρισκε η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, προβλήματα στον τομέα της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιου είδους όμως οι αντιλήψεις είναι απαράδεκτες και δυστυχώς ένα καλό άνθρωπο όπως τον νέο αυτό Ιταλό στην ουσία βλέπουμε ότι οδηγήθηκε στην δολοφονία και από θέματα τα οποία ελέγχουν μερικές φορές και αρχές άλλων χωρών. Κύριος Ντεχόσκη, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, η υπόθεση του Τζούλιο Ρετζένι πραγματικά πρέπει να θεωρηθεί αποτρόπαια και θέτει ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών μας όταν βρίσκονται στην Αίγυπτο. Ε, είναι μια χώρα, η Αίγυπτος, που θεωρούμε ότι είναι στρατικός εταίρος για το μέλλον, που είναι στο πλευρό μας, με την οποία συνεργαζόμαστε. Όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες υποθέσεις, και σε σχέση και με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο είναι πάρα πολύ μεγάλη η καταπληξή μας και το σοκ που νιώθουμε. Η Αίγυπτος Όμω, για πρώτη φορά επιτρέπει ε, ομάδα ξένων ερευνητών Ιταλών στην προκειμένη περίπτωση και βέβαια σίγουρα είναι ένα καλό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Δεν αρκεί όμω. Θέλω να καλέσω, καλέσω εκ μέρου του ΕΛΚ τη Αιγυπτικέ Αρχέ να κάνουν πάντα το δυνατόν και το παραλαμβάνω πάντα το δυνατόν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών παραγνώριζοντας εντελώς τις ε, θρησκευτικέ πεπιθήσεις, πεπιθήσεις, τι πολιτικές πεπιθήσεις. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η περίπτωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κυρία Σάκη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητή συνάδελφα, αγαπητέ Επίτροπε, θρυνούμε την απώλεια της ζωής ενός φιέστα του Ιταλού φοιτητή. Όμως ε, η βασανισμή είναι ένα συχνό φαινόμενο στην Αίγυπτο και γι' αυτό θα πρέπει να ασκήσουμε τον πιέσει ε, για την αποδοσή δικαιοσύνη αλλά και για όλες τις άλλες ε, υποθέσεις. 1.700 περιπτώσεις με βάση ΜΚΟ ε, κατά την προηγούμενη χρονιά. Είναι σαφές ότι οι αρχές επιβολής του νόμου προβαίνουν σε απαράδεκτες ενέργειες. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας Ιταλών Αιγυπτίων αλλά να είναι αποτελέσματα αποτελέσματα μιας αξιόπιστης έρευνας, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα στην Αίγυπτο και βλέπουμε ότι λιγότερο επιβάλλεται δικαιοσύνη, περισσότερο υπάρχει ατιμορρησία. Με ανησυχεί επίσης ε, η κυβέρνηση Ασίζη και η προπαγάνδα της ε, που στρέφεται επίσης κατά των αντιφρόντων, κατά των πολιτικών αντιπάλων. Το 2013 πάνω από 22.000 άνθρωποι ε, μπήκαν φυλακοί με βάση τις ίδιες Αιγυπτιακές αρχές. Καιρός πια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να υψώσει το αστημά της να ακουστεί η φωνή τους και τουλάχιστον ε, να μην ε, επιτρέψει ή διευκολύνει ακόμη περισσότερο τις ε, παραβιάσεις των δικαιωμάτων με τα προγράμματα ανταλής. Πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, οι αρχές των Αιγυπτίων και διερωτώ με ειλικρινά τα διδάγματα από το πρόσφατο παρελθόν γιατί δεν διαπνέουν και δεν καθοδηγούν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι για το 2011 τα γεγονότα και τα δάγματα θα πρέπει ακόμα να σκαθοδηγούν. Ευχαριστώ. Πέρασαν πέντε εβδομάδες από το θάνατο του Ρετζένη και κάθε εβδομάδα οι πτιακές αρχές αλλάζουν την ιστορία τους γιατί από ό,τι φαίνεται πρόκειται για μια πολιτική δολοφονία μετά από διαταγή του ε, καθεστώτος Αλσίση η κυβέρνησή μου δυστυχώς δεν βρήκε την αξιοπρέπεια να καταγγείλει αυτή την κοροϊδία και να πάλι τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται διακόπτοντας τις οικονομικές σχέσεις με το καθεστώς ε, του Αλσίζη στο όνομα υποτίθεται της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Πρόκειται για ένα δικτάτορα ο οποίος έχει σαν βασικό μέσο διακυβέρνηση στην καθημερινή τρομοκρατία. Σήμερα το Κοινοβούλιο κάνει το αξιοπρεπές, κάτι το αξιοπρεπές αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει εμείς ελευθεροκτώνα καθεστώτα όπως του Αλσίση και του Ερντογάν να τα καταγγέλουμε. Και δεν πρέπει να τους δίνουμε πόρους για να καταπιέζουν τους λαούς τους. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνο καταδικάζει τον βασανισμό και τον θάνατο του Βεντζένη αλλά ζητά να δοθούν στις Ιταλικές αρχές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να υπάρξει μια διαφανής αντικειμενική ανακριτική διαδικασία. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική της εξαφάνισης των αντιφρονούντων μετά από βασανιστήρια. Η Αίγυπτος θα πρέπει επίσης να απελευθερώσει τους κρατούμενους για λόγους ελευθερίας έκφρασης, να επιτρέψει την λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών και των ελεύθερων συνδικάτων. Στρέφομαι προς εσάς κύριε Χάν. Λέγω ότι η Αίγυπτος πράγματι είναι ένα σημαντικό εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το τίμημα πρέπει να είναι ελεγχόμενο δεν θα κλείσουμε τα μάτια λοιπόν σε αυτό το οποίο συνέβη και συμβαίνει τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος άλλος εδώ, αλλά φοβάμαι ότι ε, ε, έχουμε ένα πρόβλημα με το χρόνο στη διάθεσή μας. Ακούσαμε τους εισηγητές, ακούσαμε τους εισηγητές των πολιτικών ομάδων και θα πάμε τώρα στον συνάδελφο κύριο Πόλτσακ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει φοβερές δυσκολίες το τελευταίο διάστημα, χωρίς αυτό βέβαια να αποτελεί η αδίποτε δικαιολογία για τις παραβιάσεις από πλευρά των εκπροσωπών των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η περίπτωση του Τζούλιο Ρετζένη είναι ε, τραγική. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια θεσμοθετημένη πρακτική να ξεφορτώνονται οι κρατικές αρχές οποιονδήποτε τις ενοχλεί. Οποιονδήποτε δεν αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που έχουν ορίσει για μια χώρα σύγχρονη, όπως θέλει να είναι η Αίγυπτος, αν κρίνουμε από το Σύνταγμα του 2014 που ενέκρινε. Δεν είναι όμως σύγχρονη χώρα και οι λόγοι είναι προφανείς είναι οι αντιφάσεις μεταξύ του γράμματος και της εφαρμογής του συντάγματος. Κατοντάδες χιλιάδες ε, χιλιάδων ανθρώπων έχουν εξαφανιστεί στα χέρια των αρχών, πολλές φορές βρεθεί δολοφονημένοι. Είναι προφανές ότι δεν πληρεί τα βασικά κριτήρια για ένα δημοκρατικό καθεστώς η Αίγυπτος. Ευχαριστώ. Δημοκράτες, κύριε Ντεμόντε. Μιλάμε για ένα ψήφισμα το οποίο αφορά στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα όμως ασχολούμαστε με την υπόθεση του θανάτου του Τζούλο Ρετζένι, ένας συμπατριώτης μου ε, ερευνητής ε, με όλο το μέλλον δικό του, είχε πάει στο Κάιρο για να εμβαθύνει τις μελέτες του, αλλά δυστυχώς μετά από απερίγραπτα βασανιστήρια έχασε την ίδια του τη ζωή το Κάιρο η κυβέρνηση μας έδωσε πίσω ε, το ίδιο το σώμα του Ρετζένι αλλά δεν μας έδωσε τα στοιχεία της αλήθειας που απαιτούνται. Νομίζω ότι οφείλουμε σε αυτόν, στην οικογένειά του, στους φίλους του, και στην κοινότητα του Φιουμιτσέλο από όπου προέρχεται να πούμε την αλήθεια και ιδιαίτερα το οφείλουμε σε όλους τους νέους που πιστεύουν στην δημοκρατία, στο δικαίωμα στη ζωή το οποία κανένας δεν μπορεί να σταματήσει. Ο κύριος Μπούχνερ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα οι αρχές του κράτους δικαίου είναι κεντρικές αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει, έχουν τη θέση τους και στη στρατηγική για το εμπόριο. Πρέπει δηλαδή τις αξίες αυτές να τις στηρούν και οι εμπορικοί μας εταίροι, οι χώρες με τις οποίες αναπτύσσουμε συναλλαγές. Ωστόσο, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή παραβιάζονται, σε όλες τις χώρες δηλαδή. Ιδιαίτερα όμως για την Αίγυπτο πρέπει να πούμε ότι έχει ε, τραγικά επιδεινωθεί η κατάσταση τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο πως θέλει να απαγορεύσει αδίποτε δημόσια εκδήλωση απόψεως, ακόμη και διαδηλώσεις οι οποίες θα υποστήριζαν την κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το ψήφισμα το οποίο έχουμε να εγκρίνουμε σήμερα έρχεται την κατάλληλη στιγμή και καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατεπηγόντως να δώσει έμφαση στην ε, τήρηση των όρων που συμπεριλαμβάνουμε στις εμπορικές μας συναλλαγές με την Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ. Και παρακαλώ. Ήρθαμε εδώ για να καταδικάσουμε μία βαρβαρότητα, μία παράδεκτη δολοφονία. Είναι απαράδεκτοι οι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούν οι Αιγυπτιακές αρχές για να μην πουν την αλήθεια από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σύγκρουση εσωτερική ανάμεσα σε διαφορετικές δυνάμεις της Αιγυπτιακής κυβέρνησης. Δεν αρκεί να ζητήσουμε η κυβέρνηση αυτή να ρίξει φως. Πρέπει να σταματήσουμε αμέσως ε, τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα γεωπολιτικά και ενεργειακά συμφέροντα δεν μπορούν να δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο ο ακραίος, ε, η ακραία τρομοκρατία δεν θα πολεμηθεί μέσω της κρατικής τρομοκρατίας. Σήμερα λοιπόν συνάδελφοι δεν χρειάζεται να κάνουμε το μνημόσυνο του Τζούλιο, θα πρέπει να δράσουμε και ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί. Θέλουμε αλήθεια και δικαιοσύνη για τον Τζούλιο Ρετζένη. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λόπεθ για ένα λεπτό. Εδώ είμαστε για να καταδικάσουμε το χαμό του Τζούλη αλλά και για να θυμίσουμε πώς πέθανε όπως πολλοί ε, άλλοι ε, ακτιβιστές στην Αίγυπτο ε, πριν από πέντε χρόνια και στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Είμαστε δύο να πούμε επίση ότι στο μέλλον οι διεθνεί σχέσει και ο σεβασμός στα θύματα συνεπάγονται την αποκάλυψη της αλήθειας ε, που ε, στην περίπτωση αυτή συγκαλύπτεται. Δεν είναι απομονωμένο το περιστατικό, είναι μακρός ο κατάλογος δικηγόρων, ακτιβιστών, ανθρώπινων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων οι οποίοι ε, μπήκαν στη φυλακή και πολλοί βασανίστηκαν αλλά και δολοφονήθηκαν στην Αιγυπτό τα τελευταία χρόνια. Είμαστε εδώ για να πούμε σήμερα ότι δεν πήγε μάταιος αυτός ο θάνατος, ότι θα μα εμπνεύσει ο χαμό αυτού του νέου κατά Τρόπον ώστε σήμερα να πούμε ότι δεν ε, θα κλείσουμε πια τα ε, μάτια μας απέναντι στην αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Είναι στρατηγική όχι σχέση μας με την Αίγυπτο, αλλά η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε στις αρχές. Αιγύπτο, ευχαριστώ. Κύριος Καν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταδικάζω περίφραστα την ε, αποτρόπαιη δολοφονία του Τζούλιου Ρετζένη και εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους οικείους του. Πρέπει να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση, η οποία αποτελεί συνέχεια μια σειρά εκατοντάδων μυστηριωδών εξαφανίσεων από την ανάληψη της εξουσίας του στρατού ε, στην Αίγυπτο. Είναι πολύ όχι μόνο οι Αλοδαποί, αλλά και οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα και δεν έχουν κληθεί να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη ε, εκπρόσωποι των αρχών που έχουν ασκήσει υπερβολική βία και οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο και σε θανάτωση πολιτών. Ε, πρέπει λοιπόν να ανατραπεί αυτή η νομοθεσία η οποία οδηγεί σε μια εσωτερική καταστολή. Πρέπει η, Ευρω... η Αιγυπτιακή κυβέρνηση να πιστεί να συνεχίσει μεταρρυθμίσεις και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Αίγυπτο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι και τώρα. Ύστερα από το σύντομο αυτό κατάλογο παρεμβάσεων θα περάσουμε σε ένα μακροσκελέστερο κατά πολύ κατάλογο ε, συναδέλφων που έχουν στήσει το λόγο, που δυστυχώ όμω δεν μπορώ να οικονομήσω του πάντε για λόγου χρόνου. Κύριο Σταγιάννη έχει το λόγο. Η Αίγυπτος είναι βασικός συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντική χώρα για τη σταθερότητα στην Μεσογειακή Λεκάνη. Όμως δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τις αξίες μας να υπονομευθούν για λόγους εμπορικούς ή για λόγους πολιτικούς. Ο διάλογος με μια χώρα σαν την Αίγυπτο βασίζεται και στην απαραίτητη ε, συνεργασία ε, και στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εκτών των συνόρων της. Ε, απαιτείται περισσότερη δράση ε, και ε, από την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική δράση. Θα θέλαμε να τη δούμε πιο δραστήρια και στην, στους δύο Ιταλούς πεζοναύτες οι οποίοι κρατούνται στην Ινδία ή στην περίπτωση των δύο Ιταλών εργαζομένων που δολοφονήθηκαν στη Λιβύη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεχθήκατε και τα χειροκροτήματα των συναδέλφων. Κύριος Καπούτο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη θα πρέπει να πιέσει έτσι ώστε να αρχιθεί φως στον τραγικό θάνατο του Ρετζένη. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας δεν υπάρχει βολική αλήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό το οποίο συνέβη στον Ρετζένη θα πρέπει να γίνει γνωστό θα πρέπει η Ευρώπη να ζητηθεί να μάθουμε επιτέλους τι συνέβη στον Ρετζένη και τι γίνεται με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Είναι σημαντικός εταίρος της Ένωσης η Αίγυπτος αλλά πρέπει να σέβεται ε, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία ε, της πίστης και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το οφείλουμε στον Ρετζένη, το οφείλουμε στην αξιοπρέπειά μας. Ο κύριος Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Η δολοφονία στην Αίγυπτο του Τζούλιο Ρετζένι, ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεχύλισε το ποτήρι. Καταδικάζουμε τη δολοφονία του Τζούλιο Ρετζένι. Εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους φίλους ιταλούς συναδέλφους που πήραν πριν λίγο το λόγο. θα πρέπει η ευρωπαϊκή ένωση να στείλει ένα αποφασιστικό μήνυμα στην αίγυπτο η οποία οφείλει να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα πρέπει να αντιληφθεί η αιγυπτιακή ηγεσία ότι η καταπίεση των δημοκρατικών ελευθεριών και του αιγυπτιακού λαού αποτελεί βούτυρο στο ψωμί των τζιχαντιστών οι οποίοι καραδοκούν για να πάρουν τη ρεβάνς είναι δεδομένο ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο να εκφράσει την καταδίκη της για τη δολοφονία του τζούλιο ρετζένι. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς εκφράζω και εγώ τη βαθύτατη οδύνη μου προς τους οικείους του Ρετζένι και συμφωνώ ότι θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητη και άνευ προϋποθέσεων έρευνα του θανάτου του. Αλλά είναι μία μόνο αυτή η περίπτωση από τις εκατοντάδες χιλιάδων περιπτώσεων και θα ήθελα να καταλαβώ καλύτερα τι κάνουν οι αρχές στην Αίγυπτο. Και χτες ακόμη έγινε λόγος για την εταιρική σχέση με την Τουρκία και τα όσα πράττει ο Ερντογάν όπου θα σπεύσουμε να το απελευθερώσουμε τη θεώρηση του διαβατηρίου και να το ανοίξουμε κεφάλαια. Το ίδιο με το Καζακστάν, όταν ξέρουμε με τι κατασταλτικό καθεστώ έχουμε να κάνουμε. Και τώρα έχουμε και την Αίγυπτο. Καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό εταίρο. Αλλά επιτέλους κύριε Επίτροπε, δώστε μας κάποιους ε, οδηγούς, κάποιες ενδείξεις για το πώς θα διαμορφωθεί η σχέση μας με την Αίγυπτο στο μέλλον για να έχουμε μια καλή και ισχυρή εταιρική σχέση. Ευχαριστώ πολύ. Κούζο. Ευχαριστώ. Πριν 10 χρόνια συνδικαλίστρες από τη Μαχάλα μας ε, έδειξαν ε, ότι στην Αίγυπτο ζητείται δικαιοσύνη, ψωμί, ο Μουμπάρακ, ε, κακομαθημένος από τα τη μέλη της Ευρώπης και της ΕΠΑ. Δυστυχώς ούτε δικαιοσύνη, ούτε ψωμί, ούτε ελευθερία έφτασε στη χώρα, αλλά άλλο πραξικόπημα. Πάνω από 100 δις πληρώνει η Αίγυπτος στο στρατό και στον οποίο πουλάνε όπλα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το καθιστό έχει πάνω από 1.700 καταδίκες, θανατικές καταδίκες και έχει ε, εκτελέσει ε, εκατοντάδες ανθρώπους. Ε, ο, Τζουλιάνο, ο Τζούλιο Ρετζένι, ο οποίος βασανίστηκε φρικτά, δολοφονήθηκε όλα, όλα αυτά σε μια χώρα στρατηγικό εταίρο της Ένωσης. Δεν μπορεί να το αφήσουμε σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτό μπορεί όμως να συμβεί και το φοβάμαι πολύ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει τελικά τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το κάνει πάντα όταν τη συμφέρει και μόνο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω. Ναι. Και τώρα ο κύριος Μπονάνο, παρακαλώ. Sì, signor Presidente, io... Σε αυτή Θα ήθελα να πω ότι αν πράγματι η Ευρώπη θέλει να είναι ενωμένη, πρέπει να πει στην Αίγυπτο ή θα μας πει την αλήθεια για αυτό που συνέβη στο Ρετζένι ή αλλιώς θα μπλοκάρουμε κάθε σχέση οικονομική και διπλωματική. Αυτό θα αρκέσει έτσι ώστε να καταλάβει η Αίγυπτος ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει την οικογένεια του Ρετζένι, τον ίδιο τον Ρετζένι που δεν είναι πια ανάμεσά μας και να μην συνεχίσει να δίδει τέτοιες απαράδεκτες απαντήσεις κάθε φορά αντίθετες η μία με την άλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι εδώ η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία της Ευρώπης πρέπει εμείς να εμβαθύνουμε την έρευνα, μια έρευνα η οποία είναι ελεγχόμενη, μια έρευνα η οποία δυστυχώς δεν την χάνει των απαραίτητων εγγύησεων. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια ε, στην δολοφονία του Τζούλιο Ρετζένι. Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος έψαχνε, ε, ερευνούσε ένα σύστημα για να καταλάβει την λειτουργία του. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προσπάθειες ε, από την κυρία Μογκερίνη για να ε, μάθουμε την αλήθεια και γιατί όχι να διακόψουμε στην παρούσα φάση τις εμπορικές σχέσεις γιατί η αναζήτηση της αλήθειας είναι προτεραιότητα σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Ο κύριος Χάουιτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ως Βρετανός ε, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου εκφράζω την ε, συμπάθειά μου και τα συλληπιτήριά μου στους Ιταλούς συναδέλφους αλλά και την οικογένεια του Τζάνι Τζούλου Ρετζένι. καλώς και όλων αυτών που έχουν πέσει θύματα αντίστοιχη βίας στην Αίγυπτο. Θα παρακαλέσω τον Επίτροπο να με ρημνήσει ιδιαίτερα για τις εξαγωγές, και τη ρύθμιση των εξαγωγών εξοπλισμού παρακολουθήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις και σε επίπεδο Γερμανίας και σε επίπεδο της ομάδας των hackers που, είναι, ε, που εδρεύει στην Ιταλία. Πληροφορίες λοιπόν οι οποίες συλλέγονται και με πολύ ε, υψηλά κονδύλια για τις παρακολουθήσεις αναπτύσσει και η Αίγυπτος χωρίς καμία επαλήθευση από ανεξάρτητη αρχή ή το κοινό. Παραβαίνουν βέβαια τις αρχές των Εθνών και των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων τέτοιες ε, δράσεις και δεν πρέπει σε αυτό να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Giulio Regeni tragikus és brutális halálának körülményeit független és Ήταν βίαιος ο θάνατος ε, του Τζούλο Ρετζένη και αυτό θα πρέπει να το ερευνήσει μια αμερόληπτη ε, ερευνητική ομάδα. Φοβάμαι βέβαια ότι δεν πρόκειται να έχει άπλητο φως αυτήν την υπόθεση ποτέ. Ο νεαρός αυτό σίγουρα δεν έπεσε θύμα ενός ε, εγκλήματος του κοινού ποινικού δικαίου. Αλλά ε, αυτός ο θάνατος οφείλεται στις πολιτικές του απόψεις και στη δράση του και αυτό είναι απαράδεκτο και ακόμη και αν έγινε σε αυτή τη χώρα. Ε, Ιδίω όταν βλέπουμε ότι πέντε χρόνια μετά την Επανάσταση ε, είναι ακόμα ε, σκοτεινά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών, ίσως ακόμα πιο σκοτεινά και θολά. Η υπόθεση αυτή πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία να επαναληφθεί. Ευχαριστώ πολύ. E Αλήθεια και δικαιοσύνη για τον ρετζένι είναι το καθήκον όλων μας, αυτό πρέπει να επιδιώξουν όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι καμία οικονομική πραγματικότητα δεν θα συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες παρακολούθησης, καταστολής βασανιστήριων σε μια χώρα σαν την Αίγυπτο επανειλημμένα παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το υπενθυμίζει αυτό το κοινό μας ψηφίσμα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντιπαρατεθούμε με την κατάσταση αυτή με όλες μας τις δυνάμεις. Νομίζω ότι η περίπτωση του Ρετζένη θα πρέπει να μας οδηγήσει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει ιδιαίτερα για τους νέους που συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα και θέλουν να αλλάξει ο κόσμος. Ο Τζούλιο με τις έρευνές του ε, πλήρωσε με τη ζωή του μάλλον την έρευνα αυτή, την αναζήτηση της αλήθειας. Ugyanúgy vélekedett ebbe a kérdésben. Önél a viszont lehetősége parancsoljon. Φαντάζομαι ότι όλοι ε, καταλάβετε ότι έχουν την ίδια άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Θα σας δώσω τώρα σε εσά ε, το λόγο, πίτρο, πως Ναι, πραγματικά ε, είναι κοινή η άποψη μεταξύ όλων. Όλους μας ε, σόκαρε η ανακάλυψη της ορού του Τζούλιο Ρετζένι στο Κάιρο. Είχε εξαφανιστεί από τον Ιανουάριο, βρέθηκε νεκρός αρχές Φεβρουαρίου. Ήταν ένας νεαρός φοιτητής στο Κάιρο. Αυτή, η, αυτός όχος είναι μια προσωπική απώλεια και τραγωδία για όσους τον γνώριζαν, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα θεσμικά όργανα και για τον απλό κόσμο. Νομίζω το είπαν όλοι οι σημερινοί ομιλητέ. Η κυρία Μογκερίνη δύο φορές ε, έθεσε το ζήτημα της δολοφονίας Ρετζένη ε, στην κυβέρνηση του ΣΥΣΥ και ζήτησε να γίνει μια ανεξάρτητη ε, διαφανής έρευνα σε στενή συνεργασία με τις Ιταλικές αρχές ώστε να χειδιάπλε το φως ε, στις ε, συνθήκες του θανάτου του και για την προσαγωγή των ε, θητών, των ενόχων στην δικαιοσύνη. Υπήρξαν θεμερεί επαφέ με τι Αιγυπτιακέ αρχέ και το Φεβρουάριο. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και η ΕΕΔ παρακολουθούν ε, την υπόθεση στενή συνεργασία και συνεννόηση με την Ιταλική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία και ε, πρόθεση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε κάθε χώρα, ε, συμπεριλαμβανομένη και τη Αιγύπτου. Να σα δώσω και ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα. Είχαμε διάφορε προσπάθειε για το κλείσιμο του κέντρου Ναντίν, το οποίο ε, παρέχει θεραπευτική υποστήριξη σε θύματα βασανισμών η προστασία ε, δημοκρατίας, ε, ε, η ελευθερία, το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδης λύθη των πολιτικών στο 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση επανέν ξεκίνησε τις διμερείς της σχέσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρική σχέσης η οποία ήταν σε αναστολή από το 2010 και αυτός το κάναμε γιατί θέλαμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στον τομέα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας και να έχουμε συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος πέρυσι τον Νοέμβριο στο Κάιρο ξεκίνησε επίσης ο διάλογος για θέματα ε, πολιτικά και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά από πέντε χρόνια. Υπάρχουν στενές επαφές και με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και τις οργανώσεις και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κυρία Μογκερίνη ζήτησε πριν από τέσσερι μήνε ε, να επισκεφθεί αυτέ τι οργανώσει ε, στο Κάιρο. Επίση, με τα κράτη-μέλη, ξεργαζόμαστε μία δήλωση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην Αιγυπτό, την οποία θα εκφωνήσουμε στι 15 Μαρτίου στη Γενέβη. Οπότε και συνεδριάζει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ΕΕ. ε, Ο ειδικό απεσταλμένο των δικαιωμάτων θα επισκεφθεί τη χώρα του επόμενου μήνε, ώστε να υπάρξει συνεχής, συνεχιζόμενη συνεργασία με την Αίγυπτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε από κοινού και με τις ταλικές αρχές, ώστε να βγει στο φως η πλήρης αλήθεια και οι δράστες, για, οι υπεύθυνοι για, για το απάνθρωπο βασανιστήριο και το θάνατο του Ρετζένι να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τέτοιες απαράδεκτες τραγωδίες στο μέλλον. Συνεχίζουμε να ζητούμε ε, και να ε, επιμένουμε για την ε, η πλήρη εφαρμογή των, των, του συντάγματος του 2014 μεταρρυθμίσει στον τομέα ε, της διακυβέρνησης του κράτους δικαίου. Θέλουμε πρόοδο στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί αυτά είναι ε, προσδοκίες του ίδιου του λαού ε, της Αιγύπτου για τη σταθερότητα και για την ευημερία, την ειρήνη. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ε, στο πλαίσιο της συνεργασία μας συνεργαζόμαστε και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και τις οργανώσεις κοινωνίες των πολιτών για την αντιμετώπιση ιδίω όλων αυτών των ζητημάτων και για, την, για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Αυτός είναι και ο στόχος μας ε, γενικότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Έχουμε 8 ψηφίσματα για το θέμα αυτό και σας ενημερώνω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα μετά τις συζητήσεις μα. Τώρα έχω στην ημερήσια ένταξη τη λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό με τον κύριο Σεβαστιαν Η κατάσταση στην δημοκρατία του Κονγκό είναι σοβαρότατη. Αυτά τα οποία κάνει ο Καμπιλά για να παραμείνει στην εξουσία ενώ το εμποδίζει αυτό το σύνταγμα της χώρας του δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταστέλλονται οι διαμαρτυρίες αυτές και προκαλούν πάρα πολλά θύματα ακόμα και θανάτους. Αυτό οδηγεί στην πτωχοποίηση, την τεράστια φτώχεια που χτυπά το σύνολο του πληθυσμού της χώρας και οδηγεί επίσης και σε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο χαμηλής έντασης ανάμεσα στους πληθυσμούς του Βορρά και του Νότου και που χτυπά κυρίως τις γυναίκες. Η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων ε, υπογράφει την πρόταση αυτή για να απαιτήσει από τον Καμπυλά να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κατανοήσει ότι δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ενάντια στο Σύνταγμα και ενάντια στην βούληση του λαού. Θα πρέπει όμως να υπάρξει και μία αναφορά στο θέμα της εμπορίας των ορυκτών από ζώνες σειράξεων και συγκρούσεων δεν υπάρχει ένα εμπόριο αίματος θα έλεγα για κάποια ορυκτά, για κάποιες ορυκτές πρώτες και θα πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Ο κύριος Ντεμασμάκερ. Έχουμε φτάσει σε μία περίοδο κέρια για την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο οργανώσει των πολιτών, μη κυβερνητικέ οργανώσει, ακόμη και εταίροι του Καμπυλά ζητούν αλλαγέ και αντικατάστασή του στην εξουσία. Αλλά εκείνο επιμένει να παραμένει στην εξουσία, παρότι είναι αντίθετο αυτό με το Σύνταγμα. Η κατάσταση πολιτική επιδεινώνεται. Είναι ε, η λυγκιώδη με την οποία επιδεινώνεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει κανεί το δικαίωμα να μιλάει. Δημοσιογράφοι, οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, φυλακίζονται, δολοφονούνται, διώκονται με κάθε τρόπο. Ακόμα και νέα παιδιά ε, το Φρέγκο Μάλι θα σας αναφέρω παραδείγματα που βρίσκεται στη φυλακή πάνω από ένα χρόνο περιμένοντας την δικαστή. Πρέπει λοιπόν να διδεμαστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ουσιαστικό ρόλο για να ξεκινήσει ένας ανοιχτός διάλογος ε, για να προχωρήσει το Κονγκό, ε, να γίνει ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δημοκρατικό, που το οποίο θα συμβάλλει και στην ειρήνη που τόσο περιμένουν οι Κονγκολέζοι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράου ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η δημοκρατία του Κόγκο αντιμετωπίζει μια τεράστια πολιτική κρίση που απειλεί τη δημοκρατία. Βλέπουμε ποια είναι η απόπειρα του Καμπιλά να παρατείνει την εντολή του μέσω της καθυστέρησης της εκλογικής διαδικασίας παραβιάζοντας το Σύνταγμα και παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι μια χώρα εμβληματική της ανυπαρξίας συνοχής της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης είναι η πιο πλούσια πάντα χώρα σε επίπεδο πρώτων υλών. Βλέπουμε τις εμπορικές συναλλαγές που έχουμε με τη χώρα αυτή και θα πρέπει εμείς να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του σεβασμού των συνταγματικών ρυθμίσεων και αν θα υπάρξουν πραγματικά ελεύθερες εκλογές χωρίς παράνομη παράταση ε, της θητείας του Καμπυλά και θα πρέπει να απελευθερωθεί και ο υπεύθυνο γκοή αντιπολίτευσης για να προχωρήσει σε θεραπεία διότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο κύριος, η κυρία Γκάμπριελ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα αυτό το κατεπήγον ψήφισμα που θα συζητήσουμε την προεκλογική διαδικα... Ε, κατάσταση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Οι επόμενοι μήνε έχουν κρίσιμη σημασία και για το μέλλον τη ίδια τη χώρα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή των μεγάλων λιμνών. Ε, υπάρχουν βασικά στοιχεία λοιπόν που θέλω να τονίσω. Πρώτον, όσον αφορά τη διαδικασία την εκλογική, θέλουμε την ε, τήρηση των προποθέσεων που έχει διατυπώσει η Επιτροπή Παρατήρηση των Εκλογών του 2011 και αργότερα η επίσκεψη, ε, τα αποτελέσματα της επίσκεψης, οποίας είχα την τιμή να ηγηθώ. Χρονοδιάγραμμα για τις εκλογές, προϋπολογισμό για τις εκλογές, ε, δέσμευση για σεβασμό ε, αμελητή του συντάγματος προκειμένου να μην κυλήσει στη βία η χώρα. Δεύτερον, πρέπει να ανανεωθεί βεβαίω για λόγου ανθρωπιστικούς η παρουσία τη UNESCO και η προστασία στου πολίτε η περιφερειακή διάσταση ευρωπαϊκή αλλά και η, και η Αφρικανική Ένωση πρέπει να, να αναπτύξουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διαφυλαχθούν οι σχέσεις και να αποκλειστεί η αδίποτε περίπτωση κλιμάκωσης της βίας στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Γκέρεν. Ε, οι συνταγματικέ διατάξει ε, πρέπει να προστατεύουν ε, του πολίτε ενό κράτου από τι αυθαιρεσίε των ηθινών και σπάει η εμπιστοσύνη όταν δεν τηρούνται αυτές οι διατάξεις. Και αυτό γίνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αναβάλλονται εκλογές τάχα για να ε, τροποποιηθεί το Σύνταγμα. Ο στόχος είναι ο περχόμενος πρόεδρος να παραμείνει για τρίτη ε, θητεία. Αυτό ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε τελικά εδώ στην Ολομέλη για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Και ναι, πιστεύω ότι πρέπει. Γιατί, Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ στενά παρακολουθεί τη μεταβατική διαδικασία για Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την αρχή έχει ε, πιστεύω συνεισφέρει ε, στο να υπάρξουν απαραίτητε προποθέσει για τις εκλογές που έγιναν. Στήριξε, προσπάθησε να στήριξει τη δημοκρατία, κάτι που ζητούν και οι Κονγκολέζοι. Επομένω, το Κοινοβούλιο ε, συνεχώ πενθυμίζει στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας τι δεσμεύσει τι οποίε έχουν αναλάβει και πρέπει να τηρούν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη η κυρία Σέντρα Ροντρίγκεθ. Ευχαριστώ πολύ το ψήφισμα. Νομίζω ότι είναι ασθενές και γι' αυτό θα πρέπει ε, να εμβαθύνουμε σε κάποιες ακόμη πτυχές που ε, έχουν να κάνουν με τις καταπατήσεις των δικαιωμάτων στο Κονγκό. Πιστεύω το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να εγκρίνει μέτρα τα οποία θα θέσουν ένα τέρμα ε, στις ευθύνε των πολιεθνικών και στην χρηματοδότηση της ενόπλης σύραξης. Τον Απρίλιο του 2015 γενικός, συγγνώμη, ο Διευθυντής του Προγράμματος των Εθνών για το Περιβάλλον, έλεγε ότι το 2% των κερδών από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων ε, ουσιαστικά πηγαίνουν ε, στα χέρια των ένοπλων ε, αυτών ομάδων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν μέτρα για την αναθεώρηση και για την αποκλήση από συμβάσεις εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου δασικού και ορυκτού. Και τέλος πιστεύω θα πρέπει να μιλήσουμε ότι θα πρέπει να πάψει η αρπαγή γεών από τις πολυεθνικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρος Αρενά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Σύνταγμα του Κονγκό προβλέπει ότι πρέπει να γίνουν εκλογέ μέσα στι προσεχεί 90 ημέρε, οπότε και εκπνέει η εντολή του Πρόεδρου Καμπυλά. Ωστόσο, αυτό διατηρεί τη σιωπή του και φαίνεται ότι το σύστημα είναι διατεθειμένο να διατηρήσει την θέση του στην εξουσία. Κίνδυνο μεγάλο για τη δημοκρατία του Κόγκο. Υπάρχουν από το 2012 ιδιαίτερε πιέσει εναντίον τίποτε φωνή αντίθεση στο καθεστώ. Ζητούμε λοιπόν με το ψήφισμα πρώτον το ταχύτερο δυνατόν να εγκαθιδρυθούν οι όροι για τη διαξαγωγή ανώθευτων διαφανών και ελεύθερων εκλογών ε, η Αφρικανική Ένωση πρέπει να δραματίσει το ρόλο της, δηλαδή να κάνει σεβαστό το Σύνταγμα και τις διαδικασίες, μια διαδικασία σαφή, στοχευμένη και καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη να, να διατηρήσουν ενισχύ το, ε, την εντολή της Μενούσκο. Ευχαριστώ πολύ, Πρέντα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω στην ανάγκη διοργάνωσης ε, βουλευτικών και προεδρικών εκλογών πριν τα τέλη της χρονιάς στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα και πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή τη γραμμή να ακολουθήσουμε. Απαρέγκλητα. Ο πρόεδρος ε, Καμπιλά έχει ε, να επιλέξει μεταξύ του σεβασμού του συντάγματος άρα δύο θητείες το πολύ, και της ε, προσπάθειας να παραμείνει με κάθε τίμημα στην εξουσία. Εγώ ελπίζω να επιλέξει την πρώτη οδό, δηλαδή το σεβασμό του συντάγματος, διότι διαφορετικά φοβούμε ότι το σενάριο του Μπουρούντι και άλλων χωρών παρόμοιων θα επαναληφθεί αυτή, αυτός ο πειρασμός ε, ε, το δινικές παραμονή στην εξουσία ξέρουμε που καταλήγει. Ευχαριστώ. Κυρία Κιέγγε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι προεδρικές εκλογές στη Δημοκρατία του Κονγκό είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι μια δημοκρατική πρόκληση. Η χώρα πρέπει να αποδείξει ότι σέβεται το Σύνταγμα και τις προβλέψεις του Συντάγματος που περιορίζουν σε δύο θητείες την Προεδρία. Θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα εκλογικό με σεβασμό των αρχών του συντάγματος ζητώντας από ε, την κυβέρνηση να σεβαστεί την ελευθερία του τύπου είναι το ελάχιστο της δημοκρατίας. Ε, το τέλος λοιπόν ε, του καθεστώτος Καμπυλά είναι κάτι το απαραίτητο και θα επηρεάσει θετικά τη σταθερότητα της περιοχής ευρύτερα. Απαιτείται επίσης και η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που σέβονται το Σύνταγμα της χώρας και ζητούμε από την, από την Οργάνωση για την Αφρικανική Ενότητα να επιβλέψει την δημοκρατική μετάβαση. Ο κύριος Νάρτ, μιλώντας για την δημοκρατία του Κονγκό, είναι κάτι το ηρωνικό γιατί αυτή η δημοκρατία δεν ανήκει στο λαό, ανήκει στις ένοπλες ομάδες και στην κλεοπλεπτοκρατία είναι, υπάρχει μια μικρή μειοψηφία των, της φυλής των Μακόγκο που ελέγχει τη χώρα εις βάρος της πλειοψηφίας. Είναι κάτι το οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα αυτή στην τελευταία θέση της ανάπτυξης στον κόσμο. Έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια 100 περίπου εκατομμύρια βοήθεια ε, ε, δυστυχώς όμως δεν έχει βοηθηθεί η κοινωνία των πολιτών. Η κλεπτοκρατία εξακολουθεί να σοβεί στην συγκεκριμένη χώρα. Τα άρθρα 8, 9 και 67 ε, της Συμφωνίας του Κοτονού θα πρέπει να εξαρτήσει την βοήθειά μας προς τη χώρα με το αν η χώρα είναι πράγματι δημοκρατική. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η ασταθής ε, δημοκρατική κατάσταση και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο ουσιαστικά μας κάνει ε, να αφιβάλλουμε κατά πολύ ε, για την δυνατότητα διεξαγωγής δίκαιων εκλογών. Βλέπουμε η δυνάμεις της αστυνομίας και επιβολής της τάξης να διαλύουν με βίο τρόπο τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες και ο πρόεδρος Καμπίλα κάνει ό,τι μπορεί για να καθυστερήσει τις εκλογές και να παραμείνει στην εξουσία. Οι ε, ε, πλητοπαραγωγικοί πόροι της χώρας ε, δεν αξιοποιούνται για την ευημερία του πληθυσμού αλλά δημιουργούν διαφθορά μια νέα ε, εκλογική εφορευτική επιτροπή με μέλη από την κοινωνία των πολιτών και από την αντιπολίτευση θα πρέπει να επιβλέπει τις εκλογές του Νοεμβρίου που θα πρέπει να διεξαχθούν οπωσδήποτε τον Νοέμβριο και να είναι δίκαιες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρος είναι από το 2001 στην εξουσία, στη λαϊκή δημοκρατία του Κόγκο. Με πολύ κατασταλτικό καθεστώς, πιέσεις, βία, πρέπει να προστατευτεί το Σύνταγμα και να γίνουν εκλογές. Αν δεν συμβεί αυτό δεν μπορεί να θεωρείται μέλος της κοινωνίας των δημοκρατικών κρατών, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Είναι πλούσια σε ορυκτό πλούτο η χώρα. Αλλά δυστυχώς οι πολίτες της είναι πολύ πτυχοί. Πρέπει επίσης να συνεχίσει τις προσπαθίες του και ο οργανισμός των Αθηνών στην περιοχή υπέρ της δημοκρατίας και της ειρήνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Ε, γίνεται όμως μεγάλη οχλαγωγή στην ε, αίθουσα. Δεν έχω χρόνο, λόγω και της φασαρίας που γίνεται, να ακούσω όλους τους ομιλητές. Πετήρ, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την ανησυχία μου για την ε, πολύ σοβαρή αυτή κατάσταση στο Κονγκό. 7,5 εκατομμύρια στο Κονγκό φαίνεται ότι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό ή στην ε, νοσοκομιακή περίθλιψη αυτή τη στιγμή και πολλά είναι τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σχολείο λόγω ε, των ε, διαφόρων συγκρούσεων ε, και των στρατητικών επιχειρήσεων. Τρία εκατομμύρια είναι εκτοπισθέντες και άλλο μισό εκατομμύριο έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικέ χώρες επειδή εκδιώχθηκαν. Περιμένουμε να γίνουν οι προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο και ελπίζουμε να είναι το πρώτο βήμα προς τη δημοκρατική μετάβαση μετά από πολυετή εμφύλιο πόλεμο και πολλά χρόνια πολιτικής αστάθειας. Όλοι μαζί θα πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς στις δημοκρατικές αυτές διαδικασίες του Κόγκο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριος έχει Πρόεδρε, νομίζω ότι ο πρόεδρος Καμπιλά πρέπει να ρίξει μια ματιά γύρω του. Δυστυχώς είναι και άλλα παραδείγματα κρατών στην Αφρική αιωνίων προέδρων που προσπαθούν να απαλλαγούν από τα συντάγματά τους. Ο Πλέσταν Πορέ, παραδείγματι, στην Πορκίνα Φάσο πρόσφατα αλλά επικράτησε η βούληση του λαού και άρχισε να λειτουργεί μια δημοκρατική διαδικασία. Τα πλούτη του Κονγκό, γιατί υπάρχουν όντω, είναι πλούσια όντω η χώρα, πρέπει να κατανέμονται με βάση ένα δημοκρατικό καθεστώ στον λαό που υποφέρει τόσο πολύ σήμερα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει εταίρο τη Αφρική γιατί έχουν κοινό μέλλον και πεπρωμένο, αλλά πρέπει ταυτόχρονα και να επαγρυπνεί για το σεβασμό τη Δημοκρατία στην Αφρική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον κύριο Ντονανού. Και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση με τον Επίτροπο Χαν που θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ησυχία. Παρακαλώ, μη θορυβείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πολύ καλή η ευκαιρία συζήτησης της κατάστασης στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δημοκρατία του Κονγκό και αναμένει την αποδοχή του ψηφίσματος που ασχολείται με τις πολιτικές διαδικασίες, την πορεία προς τις εκλογές και την κατάσταση στον τομέα του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών. Η χώρα αυτή είναι μια τεράστια χώρα με τεράστιες προκλήσεις, όχι μόνο η φτώχεια, όχι μόνο η ασφάλεια, το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Μερικές φορές η χώρα αυτή μετατρέπεται οι περιοχές της τουλάχιστον σε πεδία μάχης και αντιμετωπίζει συνεχώς κρίσεις. Η εύθραυστη ειρήνη στην ανατολική πλευρά της χώρας ε, εξαρτάται από την μεγαλύτερη ειρηνευτική δύναμη. Το Μινούσκο έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ εύθραυστη ε, κατάσταση μετά από τις τελευταίες εκλογές του 2006 υπήρξε κάποια πρόοδος, η οικονομία αναπτύχθηκε, κάποιες ένοπλες ομάδες στην ανατολική πλευρά της χώρας ε, αφοπλίστηκαν και υπήρξε μία μικρή θετική εξέλιξη σε επίπεδο οργάνωσης του κράτους. Τώρα βρίσκεται σε, θα έλεγα, κρίσιμη στιγμή. Το 2016 θα έπρεπε να είναι μια χρονιά εκλογών, αλλά θεωρεί αντιπολίτευση και φοβάται ότι οι προθεσμίες οι συνταγματικές δεν θα γίνουν σεβαστές. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι εκλογές και ο δημοκρατικός τους χαρακτήρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση θα πρέπει να συμφωνήσουν σε όλα τα πολιτικά θέματα. Θα πρέπει όμως από κοινού να βρουν ένα οδικό χάρτη που να οδηγήσει ε, στην ψηφοφορία. Η δημοκρατία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ε, δυστυχώς όμως ε, οι διαμαρτυρίες οι ειρηνικές αντιμετωπίστηκαν με βίαιη καταστολή και οι δημοκρατικές ελευθερίες απειλούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας. Υπάρχουν ε, συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η δικαστική εξουσία έχει λειτουργήσει δυσανάλογα αυστηρά. Στις 8 Μαρτίου υπήρξε μια δήλωση στην Κινσάσα που υπενθύμησε στην κυβέρνηση την ανάγκη να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της. Η πρόκληση είναι τεράστια. Η οικονομία έχει θυγεί από ε, πτωτικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών και η παροχή υπηρεσιών ε, δυστυχώς ε, χειροτερεύει στην χώρα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει στην ασφάλεια, στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ανάπτυξη. Έχουμε μία μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση και θα πρέπει να βοηθήσουμε όχι μόνο σε επίπεδο υλικό, όχι μόνο να στηρίξουμε τις διπλωματικές ε, πρωτοβουλίες, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους υπόλοιπους Αφρικανούς εταίρους και τη διεθνή κοινότητα. Εμείς θέσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτα και πιο σημαντικά. Έχουμε εργαστεί στενά και με τα Ηνωμένα Έθνη ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στην ε, δημοκρατία του Κονγκό. Θέλουμε να μην υπάρχει πλέον ατιμορρησία και να τερματιστεί η σύγκρουση. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου και με τις αρχές της χώρας. Συμπερασματικά, Πρόεδρε, θεωρούμε ότι θα είναι δυνατόν η χώρα αυτά να προχωρήσει και να περάσει από την έκθραστη κατάσταση στο σεβασμό του συντάγματος στο κράτος δικαίου. Το μέλλον της δημοκρατίας του Κονγκό ανήκει κυρίως και απόλυτα στους πολίτες της. Θα πρέπει η φωνή τους να γίνει σεβαστή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να το πετύχει. Το ψήφισμα λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται σε εύθετο χρόνο και θα βοηθήσει ε, ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ και για την ειδική προσοχή που δείξατε στην ομιλία μου. Πρόεδρος, όντως και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των συναδέλφων. Όντως επικρατεί ο στην ε, αίθουσα όταν φτάνουν κάποιες εκατοντάδες συνάδελφοι ταυτόχρονα για τις ψηφοφορίες. Αυτά συμβαίνουν, δεν μπορέσαμε να σας ακούσουμε με ηρεμία και ησυχία. Έχουμε λοιπόν λάβει τα, τα σχέδια ψηφίσματος, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και όσον νούπο θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφοφορία λοιπόν.